τα συνοπτικά και τα κείμενα της χθεσινής συνεδρίασης, ε, ε, τα κείμενα που εγκρίθηκαν, ε, διατίθενται. Αν έχετε σχόλια, εάν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνονται.